Uh, Καλησπέρα σας. Δώσαμε και το ακαδημαϊκό δεκάλεπτο που έγινε δεκάλεπτο. Ας ξεκινήσουμε. Σημείο 13 στην ημερήσια διάταξη. Μείωση των ε, ε, πιστώσεων ανάληψη υποχρέωσης και των πληρωμών και θα πρότεινα αν δεν έχει αντίρρηση ο εισηγητή, τα δύο θέματα που έχει να τα συστήσουμε ταυτόχρονα. Του δίνω το λόγο. Κύριε Χάουαρντ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Το σχέδιο προπολογισμού παριθμών 4 είναι προπολογισμό που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον προπολογισμό 2019 σαν τροποποίηση με βάση και την εμπειρία που έχει από την υλοποίηση στην πράξη του προπολογισμού αυτού και έτσι κάνει κάποιες προσαρμογές στις αναλήψεις δεσμεύσεων, ε, υποχρεώσεων και τις πληρωμές. σε σχέση με την συμφωνία για τον προπολογισμό στα τέλη του 2018. Αυτές οι μεταβολές, μειώσεις ή αυξήσεις αναλόγως, μας δίνουν ένα συνολικό αποτέλεσμα μείωσης σε 100 εκατομμύρια, σε 100 εκατομμυρίων ε, ευρώ για την ανάληψη υποχρεώσεων και 50 εκατομμυρίων στις πληρωμές σε διαφορετικές ε, κατηγορίες και έτσι θα ζητήσω μετά από την Επιτροπή σας προειδοποιώ ήδη από τώρα να ετοιμαστείτε να μας εξηγήσετε λίγο ανακατηγορία το, τη λογική με την οποία μας έχετε προτείνει τις αλλαγές αυτές ώστε να καταλάβουν και οι συνάδελφοι τι πρόκειται να αντιμετωπίσουμε και να ψηφίσουμε όταν έρθει η ώρα. Από την ώρα που καταρτίστηκε το έγγραφο πρέπει να σας πω τα μέσα Ιουλίου χονδρικά έγιναν μια σειρά, υπήρξαν μια σειρά από εξελίξεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τον ε, προϋπολογισμό του 2019 προς τα τέλη του έτους. Άρα δεν θεωρώ ότι είναι η τελευταία αλλαγή στον προϋπολογισμό που θα αντιμετωπίσουμε. Οι προσαρμογές κανονικά κατατίθενται αργότερα μέσα στο έτος από τις είδαμε εμείς. Άρα ίσως να δούμε ένα άλλο σχέδιο αργότερα τροποποίησης διορθωτικού προπολογισμού δηλαδή. Αυτή λοιπόν η σημαντική προσαρμογή και διόρθωση στην οποία αναφέρομαι κατά πάσα πιθανότητα θα επηρεαστεί και από τη διαδικασία δυστυχώς του Brexit είναι πιθανόν και το πολιτικό σενάριο στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει μετατοπιστεί από την ώρα που είχε σταχθεί το έγγραφο για το οποίο συζητούμε. Είναι πιθανόν λοιπόν η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στον προπολογισμό Εάν μπορούμε βέβαια να πιστέψουμε τα όσα λέει η Βρετανική κυβέρνηση και αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι εύκολο κάτι τέτοιο για όλους, ε, θα οδηγούσε σε μια ευνίδια αποχώρηση από 1η Νοεμβρίου και άρα ε, πάυση συμβολή στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό του Ηνωμένου Βασιλείου στην, στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα το οποίο βεβαίως θα επηρέαζε και τον προπολογισμό συνολικά. Ε, από τα όσα θα έχετε διαβάσει στον τύπο τις τελευταίες ημέρες, θα παρατηρήσατε φαντάζομαι ότι έγινε μια συνάντηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τετάρτη με μια συζήτηση για την τροποποίηση της νομοθεσίας που αφορά το Ταμείο Αλληλεγγύης, πράγμα το οποίο θα ήταν σημαντικό ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που θα α, αντιμετώπιζαν οι πιο ευάλωτες περιοχές Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση άτακτου Brexit. Αυτά τα είδαμε και στο Ρωμανό Βασίλειο, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δημοσιεύονται. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο βεβαίω θα ήταν κάπως παράλογο να μειωθεί αυτή τη στιγμή σε αυτή τη χρονική περίοδο το Ταμείο Αλληλεγγύης. Πάντως θα ήθελα να σας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πληροφορίες και περιμένω να ακούσω τι ε, θεωρούν οι συνάδελφοι από τις άλλες ομάδες ότι θα πρέπει να γίνει. Εγώ θα έλεγα κλείνοντας και τη βλέπω να υπάρχει μια σύμπτωση στα οικονομικά στοιχεία ότι κάθε σχέδιο προπολογισμού είναι διαφορετικό από τα άλλα. Ωστόσο εδώ βλέπουμε συνολικά ποσά για να σας διευκολύνουμε και όπως είπα, ανάλογα με το τι έκβαση θα έχει αυτός ο διορθωτικός προϋπολογισμός, το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού, μπορεί να γίνουν κάποιες άλλες ε, συζητήσεις στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θα ακούσουμε τώρα τους κοιόδης ηγητές ε, με την κυρία Χολμάια. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ λίγο πολύ στα ίδια θα σταθώ και προς την ίδια κατεύθυνση με τον συνάδελφο στον ΤΑΠ 4 παραδείγματι βλέπω πως είναι όλο τυχαίο το ότι 100 εκατομμύρια σε άλλο ε, ε, σε άλλη γραμμή του προπολογισμού βγαίνουν, σε άλλη κατηγορία μάλλον βγαίνουν, ενώ σε άλλη προστίθενται. Ενδιαφέρον να το κοιτάξουμε λίγο πιο προσεκτικά. Και μάλιστα σε κάποια επιμέρους σημεία πρέπει να πω πως με ευνηδιάζει το γεγονός ότι με κάποιες μειώσεις καταφέρνουμε τελικά να τα βγάλουμε πέρα. Στο δε σημείο Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας θα ήθελα να ξέρω γιατί ξαφνικά χρειάζονται τόσο πολλά λιγότερα χρήματα. Είμαι βέβαιη ότι δεν έχουν καμία σχέση αυτά με τον DAB 2 και θα ήθελα να μου δώσετε κάποια εξήγηση. Η κυρία Αχμό έχει το λόγο. Κατανοώ πως κανείς θέλει να προλαβαίνει το τέλος της χρονιάς, αλλά πιστεύω πως είναι λίγο νωρίς ακόμα. Αν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ζητά να απελευθερώσουμε αυτά τα 100 εκατομμύρια, και είναι ένα θέμα το οποίο θίξαμε και σήμερα το πρωί. Ε, έχουμε τη Γενική Εισαγγελία, αν μας περισσεύουν κάποια χρήματα να τα προσθέσουμε εκεί, λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά. Αλλά αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί μια περικοπή 100 εκατομμυρίων, τι σημαίνει ότι αυτά είναι πια διαθέσιμα για να τα πληρώσουμε κάπου αλλού. Ε, να τα τοποθετήσουμε στην άκρη για άλλες ανάγκες. Τι πιστεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πως σε κάποια θέματα πρέπει να τα κοιτάξουμε από πιο κοντά. Ναι, ίσως έχει δίκιο. Ίσως χρειαζόμαστε σε κάποιες περιπτώσεις λιγότερο χρήματα. Αλλά καλό θα ήταν να μας τα εξηγήσουν έτσι ώστε να έχουμε και ένα περιθώριο κινήσεων ε, σε κάποιους άλλους τομείς, μια και έχουμε 4-5 μήνες μπροστά μας μέχρι το τέλος της χρονιάς και καλό θα ήταν να έχουμε αυτή την ελευθερία ελιγμών. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Άντρες. Δεν έχουμε πολλά να προσθέσουμε. Νομίζω τα πιο σημαντικά έχουν ήδη υποθεί από άλλους. Τους στηρίζουμε. Έχουμε κάποιες τεχνικές προσαρμογές που είναι απαραίτητες και να σας πω πως έχω πάρα πολλές ερωτήσεις σχετικά με κάτι που συζητάμε ε, για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό ε, πλαίσιο και για τις επιστροφές που λαμβάνουν κάποια κράτη-μέλη. Αλλά νομίζω θα έχουμε το χρόνο και θα το συζητήσουμε αργότερα όταν μιλήσουμε για το θέμα των ε, δημοσιονομικών ε, προοπτικών. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα κι εγώ να κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις και να σας πω πως εμείς ως ομάδα στηρίζουμε ε, τα όσα συζητήσαμε ε, προηγουμένως. Άρα ναι, εμείς είμαστε υπέρ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας δώσω κάποιες σύντομες εξήγησει για να δείτε τι έχουμε σε αυτό το σχέδιο ε, προσαρμοσμένου προϋπολογισμού. Οι τροποποιήσεις λοιπόν αυτές είναι κάποιες προσαρμογές που έγιναν μέσα στη χρονιά για να λάβουν υπόψη και τον ρυθμό εφαρμογής και εκμεταλλεύσεων και επίσης τις ε, διάφορες εξελίξεις στις ε, νομικές διαδικασίες και τις προσαρμογές που χρειάζονται στα τελικά ποσά που συμπεριλαμβάνονται στον ευρωϊκό προϋπολογισμό. Για το κομμάτι των δαπανών, να σας πω πως έχουμε από μία, σειρά προσαρμογών, μία μείωση δηλαδή 18,5 εκατομμύρια ευρώ για τις ε, Ευρωπαϊκές Αρχές ε, Εποπτείας και αυτό έχει να κάνει με το τελικό αποτέλεσμα της νομικής διαδικασίας για τις τρεις αυτές εποπτικές αρχές όπου το ποσό που τελικά απαιτείται είναι χαμηλότερο από αυτό το οποίο είχε προβλεφθεί αρχικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το οποίο είχε ε, συμπληρωθεί στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 19-20. Αυτό λοιπόν είχε να κάνει με προσαρμογές ε, λόγω νομικής διαδικασίας Frontex και εκεί έχουμε μια μείωση 12 εκατομμύρια γιατί η θέση εφαρμογή της νέας νομικής βάσης, βάσης της Frontex έλαβε χώρα αργότερα από ό,τι είχε προβλεφθεί. Όταν δηλαδή ετοιμάζαμε το σχέδιο οικονομισμού για το 2019 και η δυνατότητα προσλήψεων για τη Frontex ξεκίνησε αργότερα από ό,τι είχε προβληθεί πέρσι, οπότε όλα αυτά έχουν προσαρμοστεί σε αυτά τα οποία είναι λογικά να γίνουν ε, σε επίπεδο προλήψεων ε, στην Frontex μέχρι να κλείσει το 2019. Αυτό ισχύει και για το αποθεματικό που είχαμε στον προπολογισμό του 2019 για το Δουβλίνο το οποίο επρόκειτο να ε, χρησιμοποιήσουμε για να καλύψουμε έκτακτες ανάγκες. Ένα κομμάτι έχει χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια ε, των, ε, της χρονιάς στα πλαίσια κάποιων μεταφορών με τις οποίες συμφώνησε και η Επιτροπή σας. το ποσό που έχουμε στη διάθεσή μα στο αποθυματικό είναι παραπάνω από αυτό το οποίο θα χρήσουμε μέχρι τα τέλη της χρονιάς, οπότε και εδώ έχουμε μία μείωση η οποία είναι κάτι παραπάνω από 7 εκατομμύρια. Για το πρόγραμμα Rescue, και εδώ είχαμε και συγκεκριμένη ερώτηση. Δεύτερη χρονιά έχει προσαρμοστεί το ποσό σε αυτό το οποίο συμφωνήθηκε μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, νομική βάση. Άρα λοιπόν για το 2019 η μείωση μας φέρνει στο συμφωνηθέν ποσό για το 2019 και δεδομένων των αναγκών μέχρι τα τέλη της χρονιάς πιστεύουμε πως το ποσό που βλέπετε είναι αρκετό για τις ανάγκες που καλύπτει το πρόγραμμα Rescue. Η μείωση εδώ είναι της τάξης του 35 εκατομμυρίων. Ταμείο Λιλεγγύης αυτό σχετίζεται με τα διαθέσιμα ποσά ως προκαταβολές στον ετήσιο προπολογισμό, γιατί μπορεί να χρησιμοποιήσει κανεί τι προκαταβολές έτσι ώστε να χρηματοδοτήσει κάποιε ανάγκε στα πλαίσια φυσικών καταστροφών ή άλλων καταστροφών, εφόσον έχουν κριθεί επιλέξιμες, ε, επιλέξιμα τα αιτήματα των καρτών μελών. Μία σχεδόν 30 εκατομμύρια ευρώ και εδώ. Γιατί, Γιατί είχαμε μεταφορά ποσού carry over από το 18 στο 19 εκεί είχαμε αυτή τη μεταφορά των 29,5 εκατομμυρίων ευρώ που είναι διαθέσιμα για το 19 και για τις ε, προκαταβολές στον ετήσιο προϋπολογισμό είναι 50 εκατομμύρια. Έχουμε εκεί ακόμα τα 50 ε, εκατομμύρια άθικτα, οπότε αφαιρούμε ε, τα 29,5 και έτσι λοιπόν έχουμε το απαραίτητο ποσό για προκαταβολές μέχρι τα τέλη της χρονιάς και εκεί. Δαπάνες. Έχουμε και κάποιες αυξήσεις. Γιατί, γιατί είχαμε μία καθυστέρηση στην ημερομηνία του Brexit που είχε προβληθεί να είναι νωρίτερα φέτος και όχι 31 Οκτωβρίου. Έχουμε τρία θεσμικά όργανα που έχουν ζητήσει να αυξήσουμε τις ε, ε, αναλήψεις υποχρεώσεων για δαπάνες τις οποίες είχαν πιστέψει ότι θα εξοικονομήσουν είναι το ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ελεγκτικό Συνέδριο και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Αυτά λοιπόν τα προσθέτουμε στον πολογισμό και τα είπε και ο εισηγητής με καθαρές δεσμεύσεις ε, που οδηγούν σε μία μείωση των 100 εκατομμυρίων ευρώ αν κάνουμε προς το αφαίρεση ε, ε, των ποσών που έχουμε στις πληρωμές και να σας πω που και στα έσοδα έχουμε κάποιες προσαρμογές όπου έχουμε λάβει υπόψη και, και την ε, βάση του ε, ΦΠΑ ε, που έχουμε τα έσοδα από την Τελωνιακή Ένωση αλλά και τα στοιχεία από το GNI λαμβάνοντας υπόψη και κάποια στοιχεία τι εμπορικέ ροέ και για τους ίδιους πόρου και τις συνεισφορές των κρατών μελών έχουμε εδώ κάποιες μικρές αλλαγέ για, την... για ολόκληρο το έτος. Το επίπεδο των συνεισφορών δεν αλλάζει σφαιρικά, αυτό άλλωστε ορίζεται από τον προϋπολογισμό, αλλά γίνεται μια αναδιανομία ε, ανάμεσα στα κράτη-μέλη για να ενημερώσουμε, ε, λαμβάνοντας υπόψη και τις πιο πρόσφατες οικονομικές ε, πληροφορίες. Επίσης, προς ενημέρωση, να σας πω πως ξέρουμε πως το Συμβούλιο στην Κορεπέρ ενέκρινε αυτό το σχέδιο τροποποιητικό προϋπολογισμού και ελπίζω πως σύντομα θα κάνει κάτι το αντίστοιχο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε να ρυθμίσουμε τον τρέχοντα προϋπολογισμό ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που έχουμε μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε άλλα σχόλια. So I give the word to Mr. Howard to conclude. κύριος Χάουαρ τότε για να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Οι πληροφορίες ε, που μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που ουσιαστικά περιλαμβάνονται και στα έγγραφα φαντάζομαι ότι μας δίνουν τροφή για σκέψη σε ό,τι αφορά το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού. Και θα περιμένω από πλευρά σα, από τι της τροπολογία. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Άρα, ολοκληρώνεται τα σημεία 13 και 14 τη διάταξη και θα ήθελα να σα υπενθυμίσω εδώ ότι 6 Σεπτεμβρίου, 10, λίγη, 10 η ώρα, λίγη προθεσμία για την κατά τροπολογιών ε, για το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού υπαριθμών 4 και για την απόφαση περί τροποποίησης, δηλαδή της απόφασης για το μηχανισμό ευελιξίας. Και περνάμε στο επόμενο σημείο της μέσης διάταξης, κτηριακή πολιτική. Λάβαμε μία έγκαιρη προειδοποίηση για δύο ε, κτηριακά έργα, για το EU Λίσα το ένα και για το, το δεύτερο. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Κέλλερ που είναι η μόνιμη εισηγήτρια για αυτά τα θέματα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Το πρώτο θέμα αφορά την επέκταση του κτηρίου του οργανισμού Ήγιου e που έχει έδρα στο Ταλίν και επιχειρησιακό κέντρο, δηλαδή κέντρο διαχείρισης δεδομένων των αρχείων στο Στρασβούργο. Επίσης έχει εκπροσώπηση στις Βρυξέλλες. Νομίζω ότι η ε, πρέπει να είναι και εδώ στην αίθουσα σήμερα. Ορίστε, πίσω εκεί είναι η κυρία. Ο οργανισμός EU πριν από κάποια χρόνια γνώρισε μια φάση ανάπτυξη, αλλά σε ό,τι αφορά την αποστολή της ε, και το έργο που έχει αναλάβει για σημαντικά ζητήματα όπως είναι το σύστημα εισόδων-εξόδων, το σύστημα πληροφοριών που αφορά το Eurodac και την αναδιατύπωση για το Eurodac και το σύστημα θεωρήσεων διαβατηρίου ETIAS που είναι σε εξέλιξη, το ευρωπαϊκό ΕΣΤΑ. Για όλα αυτά απαιτείται μια συμπληρωματική αναδιάρθρωση του οργανισμού που θα προέβλεπαν και σημαντική αύξηση του προσωπικού και για τεχνικά ζητήματα μεταξύ άλλων και για θέματα διαλειτουργικότητας και επικοινωνίας, δηλαδή μεταξύ των διαφόρων αρχείων για την ανταλλαγή και τη στάβρωση πληροφοριών. Κάτι πολύ σημαντικό. Για όλους αυτούς τους λόγους υπάρχει υπομελέτη ένα σχέδιο για 7.500 τετραγωνικά μέτρα θα το έχουμε με περισσότερες λεπτομέρειες στα μέσα της επόμενης χρονιάς και τα έργα κατασκευής αναμένεται να ξεκινήσουν το 2021. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, κάποια σχόλια, μήπως ερωτήσεις. Συλένθιο. Υπάρχει ησυχία, ηρεμία. Άρα κλείνει αυτό το σημείο, γιατί δεν υπάρχουν σχόλια, απλά να πω ότι ξεκολουθούμε να περιμένουμε τα ονόματα των σχεδόν εισηγητών για τα κτίρια και ελπίζω να τα έχουμε σύντομα. Παρακαλώ να το λάβετε υπόψη σας οι πολιτικές ομάδες. Σας ευχαριστώ. Ξέχασα το δεύτερο, το EAS, δηλαδή την ΕΙΕΔ, την Υπηρεσία εξωτερική Δράσης. Δεν μιλήσατε, κυρία Κέλλερ, για την ΕΙΕΔ. Α, πήγα πολύ γρήγορα. Ναι, πράγματι υπάρχει το δεύτερο project, η ίδια υπηρεσία με αυτή που αναφέραμε το πρωί, ε, που είναι υπηρεσία εξωτερικών σχέσεων. Για αυτή την υπηρεσία απαιτούνται παρεραιτέρω κτίρια, διότι με βάση και το project το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί αφορούσε το προσωπικό όπως είχε οριστεί πριν απο δυο δύο-τρία χρόνια και οι παρόντες συνάλλευοι ενέκριναν αύξηση 46 ισοδύναμων θέσεων για τον προπολογισμό του 2019, αύξηση προσωπικού λοιπόν, για την οποία όπως καταλαβαίνετε απαιτεί ούτε 3 με 4 χιλιάδες επιπλέον τετραγωνικά μέτρα, έκταση, επιφάνεια για τα γραφεία αυτά. Έχουν ξεκινήσει σχετικές εργασίες και για την πρόσληψη του πλέον αυτού προσωπικού. Είπαμε ότι ζητούμε αύξηση του προπολογισμού 5 εκατομμύρια για θέματα ασφάλειας κυρίως. Δεν ε, προβλέπεται όμως ε, γι' αυτό. Γι' αυτό και θέλουμε να ληφθεί υπόψη ε, πλέον του ότι αποφασίσαμε το πρωί. Αλλά επειδή νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι χρειάζεται αυτή η στελέχωση και, και η κτηριακή αυτή υποδομή. Νομίζω ότι πρέπει να τύχει ευνοϊκής μεταχείρισης αυτό το έργο. Ευχαριστώ. Ναι, συγγνώμη, εγώ φταίω που δεν θυμήθηκα να σας δώσω το λόγο και για το δεύτερο project. Υπάρχουν ερωτήσεις, λέει ο πρόεδρος. Όχι. Και τώρα κλείνω την σημερινή συνεδρίαση, παραλαμβάνοντα ότι χρειάζομαι τα ονόματα των σχεδόν εισηγητών για τα κτίρια επόμενη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες ε, στις 23 και στις 24 Σεπτεμβρίου.